και είπατε εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας για την εκλογική διαδικασία στην ΑΙΤ. Από πλευράς της Επιτροπής και εκπροσωπώντας την Αντιπρόεδρο καλωσορίζουμε την Επίτροπο Κρέτου η οποία και έχει το λόγο. So, uh, dear uh, Αγαπητή Πρόεδρε, Κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη, από πλευρά τη υπάτη εκπροσώπου, Χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να είμαι σήμερα μαζί σα να συζητήσουμε την ΑΕΤ και τη σοβαρή πολιτική και θεσμική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα. Η κατάσταση τη προκαλεί πολλή ανησυχία και είναι πλήρως αιτιολογημένο να αντιμετωπίσουμε σήμερα αυτό το θέμα. Η πρόσφατη αναβολή επαόριστον του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών που αρχικά προβλέπονταν για τις 27 Δεκεμβρίου και κατόπιν για τις 24 Ιανουαρίου έχει προκαλέσει μια περίοδο ανασφάλειας και τον κίνδυνο ενός θεσμικού κενού Άρα ο λαός της μπορεί να μην μπορέσει να ασκήσει πλήρως το δημοκρατικό δικαίωμα να εκλέγει τους αρχηγούς του. Και επειδή υπάρχει γενικά έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς και χαμηλή συμμετοχή σε εκλογές, η προετοιμασία του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών έγινε σε ένα ιδιαίτερα πολλωμένο περιβάλλον με κατηγορίες νοθείας από πολλούς συμμετέχοντες. Η προσωρινή εκλογική επιτροπή είδε διάφορα μέλη της να παρετούνται και η κλιμάκωση της βίας έχει ήδη προκαλέσει πολλούς θανάτους και γι' αυτό αποφάσισε η Επιτροπή αυτή να αναβάλει τις εκλογές. Και η κατάσταση αυτή, ιδιαίτερα σε μια χώρα σαν την Αϊτή, όπου υπάρχει πολύ εκτεταμένη φτώχεια και πολλά ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Αυτή η κρίση μπορεί να θέσει εν κινδύνο τις προσπάθειες ανοικοδόμησης και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μετά τις τρομερές καταστροφές του σεισμού του 2010. Τα αποτελέσματα αυτά στην ανοικοδόμηση επετέφθησαν λόγω στην ε, μεγάλη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ε, ανοικοδόμηση της χώρας. Στείλαμε τον περασμένο Ιούλιο μια πολυμερή αντιπροσωπεία παρατήρηση των εκλογών με επικεφαλή στην κυρία Βαλενθιάνο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αποτείω φορό τιμή στην ε, συμβολή τους έδωσαν μια ανεκτήμητη υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ΑΕΤ χάρη στον ευσυνείδητο και ανεξάρτητο τρόπο με τον οποίο παρατήρησαν τις εκλογές. Η αποστολή αυτή ανέφερε ότι υπήρξαν διάφορες παρατυπίες αλλά κατέληξε ότι δεν είχε υπάρξει μαζική νοθεία στις εκλογές τη 25 η Οκτωβρίου και ότι κατά συνέπεια το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου όπω ανακοινώθηκε ήταν σε μεγάλο βαθμό σωστό. Δυστυχώς όμως οι υποψήφοι που δεν ήρθαν πρώτοι στον πρώτο γύρο των προεδρικών αυτών εκλογών αρνήθηκαν να αποδεχθούν το αποτέλεσμα αυτών. Έκαναν αβάσιμες ε, κατηγορίες ότι υπήρξε μαζική νοθεία και έτσι μειώθηκε η εμπιστοσύνη του πληθυσμού στην διαδικασία και οδηγηθήκαμε σε αυτό το αδιέξοδο. Οι εκλογοί σίγουρα δεν μπόρεσαν να ασκήσουν πλήρως τα εκλογικά τους δικαιώματα. Κατά συνέπεια, δεν θα υπάρξει εκλεγμένο πρόεδρος μέχρι τι 7 Φεβρουαρίου. Οπότε, σύμφωνα με το Σύνταγμα, ο πρόεδρος Μαρτέλη θα πρέπει να εγκαταλείψει το αξιωμά του. Το Σύνταγμα δεν ε, προβλέπει επακριβώς τι θα γίνει, αλλά περιέχει διατάξεις για περιπτώσεις που δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του ο πρόεδρος και γίνονται διαπραγματεύσει στην ΑΕΤ αυτή τη στιγμή. Όλοι παρακολουθούμε τι εξελίξει, πολύ εκ του σύνεγγης. Ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών και η Ειδική Αποστολή Διαμεσολάβησης και μια παρόμοια αποστολή της Επιτροπής Κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής προβλέπεται να πάνε. Ελπίζουμε να προκύψει μια γενική συνένεση για να ολοκληρωθεί σύντομα η εκλογική διαδικασία με βάση την εκφρασμένη βούληση του λαού της ΑΕΤ και ελπίζουμε να υπάρξουν βελτιώσεις διαδικασία. Η αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί επίσης να συμβάλλει ιδιαίτερα. Ωστόσο, υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί συμφωνία βράχη πρόθεσμα και ότι η προσωρινή κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει θέματα νομιμοποίησης. Αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη δημοκρασία και για τη χώρα. Για δημοκρατία, για τη χώρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μακροπρόθεσμα δεσμευμένος εταίρος της ΑΕΤ σε αυτές τις δυσχερείς περιστάσεις καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν κάθε εκδήλωση βίας και να αναλάβουν τις πολιτικές δημοκρατικές τους ευθύνες. Η δημοκρατία είναι αναγκαία για βιώσιμη ανάπτυξη. Και προσβλέπω στη συζήτηση και στις απόψεις που θα εκφράσετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ κύριε Επιτρόπε. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Πρώτος είναι ο κύριο Στία. Δύο Κυρία Πρόεδρε, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Βαλενσιάνο και όλους τους άλλους ε, συναδέλφους που συμμετείχαν ε, στην εκλογική αποστολή στην ΑΕΤ. Και διαπίστωσαν το τι έγινε με τις εκλογές συνέβαλαν στην εκλογική διαδικασία. Ε, διαπίστωσαν πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της ε, εκλογικής διαδικασίας και αυτό βέβαια δεν εκπλήσει. Δεν εκπλήσει λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται αυτό το κράτος Καραϊβικής. Διαπίστωσαν όμως ότι οι εκλογές ήταν ανώθευτες, αδιάβλητες, ότι έγινε σεβαστό το αποτέλεσμα των εκλογών από το λαό της Αιτής. Πιστεύω ότι οποιαδήποτε άλλη άποψη θα ήταν απαράδεκτη. Πάντως το ΕΛΚ πιστεύει ότι πρέπει να δεχτούμε το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των εκλογών και το συντομότερο δυνατόν να ακολουθήσει ο δεύτερος γύρος έτσι ώστε η τι να έχει ένα πρόεδρο που θα διαδεχτεί τον ε, πρόεδρο Μαρτελή. Ε, όλα τα πολιτικά κόμματα οφείλουν να συμβάλλουν στην ε, ηρεμία σε αυτή τη χώρα, κάτι που είναι απολύτως απαραίτητο γιατί στις 7 Φεβρουαρίου εκπνέει η εντολή του Πρόεδρου. Η ΑΕΤ είναι μία από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου. Το 2010 η κατάσταση επιδεινώθηκε λόγω του σεισμού και ως εκ τούτου δεν είναι καλό να υπάρχει κενό εξουσίας στη χώρα. Δημοκρατική πρέπει να είναι η μετάβαση και να γίνουν προσπάθειες για να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια. Η κυρία ε, Βαλέντσια. Η κυρία Βαλεντσιάνο. Το πρώτο το οποίο θα ήθελα να κάνω είναι να επιβεβαίωσω την ευρωπαϊκή δέσμευση ενώπιον του λαού της ΑΕΤ και των ε, συνταγματικών αρχών της μια ευρωπαϊκή δέσμευση την οποία μεταφράζουμε σε αλληλεγγύη προς τους ε, πολίτες ε, της χώρας αυτής από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τα όσα βίωσε. Επομένως η πρώτη μας δέσμευση ε, με την IT είναι αυτή. Δεύτερον, θα ήθελα να πω ότι είχα την τιμή, έχω την τιμή ε, να ηγούμε μια ομάδα ε, εγνωσμένου κύρου ε, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα δημοκρατία ανά τον κόσμο και έκαναν εξαιρετική δουλειά στην παρακολούθηση τη εκλογική διαδικασία που δυστυχώ έχει παρεκτραπεί προ το παρόν στην ΑΕΤ. Η εργασία ήταν πολύ σοβαρή, ε, επισταμένη και πραγματικά όλοι οι συνάδελφοι μπορούν να είναι ήσυχοι και αν δεν είναι μπορείτε να συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα μας και τις εκθέσεις για να διαπιστώσετε ότι έχουμε τη δυνατότητα να επιβεβαιώσουμε ότι οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου που ήταν ο πρώτος εκλογικός γύρος στην αιτή ήταν σίγουρα οι πιο ε, καθαρές και λιγότερο βίαιες εκλογές που έχει βιώσει η ΑΕΤ στην ιστορία της. Και επίσης επιβεβαιώνουμε ότι τα αποτελέσματα αυτών των εκλογών στον πρώτο γύρο θα μπορούσαν ίσως ε, να οδηγήσουν ε, στο, σε ένα δεύτερο γύρο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει συνταγματική κρίση, ε, θεσμική κρίση στην ΑΕΤ, υπάρχει ένα διέξοδο το οποίο πρέπει να επιλύσουν οι ΑΕΤΙΝοί. Οι αρχές της ΑΕΤ και ο λαός της ΑΕΤ είναι αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να επιλύσουν αυτή την, το σημαντικό αδιέξοδο. Ε, το οποίο ανέλησε εξαιρετικά η κυρία Κρέτσου και εγώ δεν θα ήθελα να ε, ε, επιμείνω. Μακάρι να μπορέσουν να επιλύσουν το αδιέξοδο μέσω διαλόγου και συνένεσης. Αλλά η σύστασή μας, η ταπεινή μας γνώμη βάσει ε, σοβαρής, αυστηρής και δεσμευμένης εργασίας είναι να γίνει ο δεύτερος γύρος των εκλογών στην ΑΕΤ. Θα ήταν το πιο λογικό. Περιμένουμε λοιπόν τη λύση που θα μας δώσουν οι Αττινοί και αν πραγματικά υπάρξει δεύτερος γύρος η αποστολή παρατήρηση των εκλογών θα είναι παρούσα για να δώσει την ε, ε, επιβεβαίωσή της στη μαρτυρία της. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπιλτμπάου Μπαραντίκα στη συνέχεια για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Επίτροπο. Πριν ε, ξεκινήσω με την παρέμβασή μου θα ήθελα να ευχαριστήσω και την ομάδα η οποία εργάστηκε και στην ΑΕΤ και για την εκπόνηση της έκθεσης αλλά και την Έλενα Βαλενθιάνο για τη δουλειά της και για τη συνεργασία της και τον συντονιστικό ρόλο που ανέλαβε με αυτή την ομάδα του Κοινοβουλίου. Ως ε, υπεύθυνη της αποστολής παρατήρησης ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου νομίζω ότι το βασικό μας καθήκον από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων είναι να ζητήσουμε να γίνει ο δεύτερος γύρος ο οποίος αναβλήθηκε στις 24 ε, Ιανουαρίου για πολλωστή φορά για να μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά σε ένα δεύτερο γύρο. Η ολοκλήρωση αυτής της εκλογικής διαδικασίας είναι ο καλύτερος τρόπος να ε, ε, μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την ε, κρίση που δημιουργείται από την αποχώρηση του κυρίου Μαρτελή και να υπάρχει ένας νέος πρόεδρος στην ΑΕΤ. Ο πρώτος γύρος έγινε με ηρεμία, χωρίς τα περιστατικά βίας που είχαμε στις 9 Αυγούστου. Επιτόπου διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν προβλήματα όπως ε, μικρή συμμετοχή, κάποια διάκριση ίσως στην υποβολή των υποψηφιωτήτων και κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να βελτιωθούν όσον αφορά τις κυρώσεις για όσους ήταν υπεύθυνοι για τις βιαιότητες ε, στις προηγούμενες εκλογές. Αλλά την ημέρα των εκλογών υπήρχαν πολύ σημαντικές πρόοδοι για τη δημοκρατική ε, νοοτροπία της χώρας. Πρόκειται για μια από τις φτωχότερες χώρες του πλανήτη και οι κάτοικοι της ε, αξίζουν να εγκαταλείψουν αυτή την οικονομία της υποστήριξης και του πόνου και να μπορέσουν να ξεπεράσουν αυτή την ιστορία της καταπίεσης και της βίας. Επομένως ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποια πράγματα για αυτές τις κοινωνίες οι οποίες προσπαθούν να προχωρήσουν και να μπορέσουμε να καταλήξουμε στο διάλογο και στο κράτος δικαίου. Η ΑΕΤ χρειάζεται λόγους για να πιστέψουν ότι αυτοί κρατούν στα χέρια τους το μέλλον τους και οι εκλογές ε, ε, χρειάζονται για κάποιο λόγο. Κάποια παιδιά μας κοιτούσαν έκπληκτα, οι ενήλικες προσπαθούσαν να βρουν μια ελπίδα ε, σε αυτές τις εκλογές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από μεγάλη αβεβαιότητα και βρίσκονται σε κατάσταση πολύ μεγάλης φτώχειας, επομένως τους αξίζουν δημοκρατικά θεσμικά όργανα για να μπορέσουν να έχουν ευημερία στο μέλλον και ένας τρόπος να το επιτύχουν αυτό είναι να μπορέσουν να εκλέξουν δημοκρατικά ένα νέο πρόεδρο, τον οποίο θα νιώθουν ότι είναι δικό του άνθρωπο, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το κράτο δικαίου και να έχουμε και τι ε, ε, συνενέσει που χρειάζεται η χώρα για να προχωρήσει. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Βριζιά. 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών αναβλήθηκε εκ νέου. Το πολιτικό αδιέξοδο στην ΑΕΤ είναι ανησυχητικό. Δεν θα σας κόβουμε όμως να δραματοποιούμε την κατάσταση υπερβολικά. Η οικοδόμηση μιας σταθερής δημοκρατίας ε, δεν είναι κάτι εύκολο και ξεκινάει από πολύ χαμηλά η ΑΕΤ. Συμμετείχα στην αποστολή, ευχαριστώ όλους που ήταν μαζί μας. Παρατήρησα ότι οι ΑΕΤιανοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την διαδικασία και τους πολιτικούς ηγέτες. Αυτό το αποδεικνύει και η υψηλή αποχή πάνω από 90%. Είναι επιτακτικό να αντιμετωπίσουμε τα βαθιά αίτια αυτής της δυσαρέσκειας. Φασίζεται στη μία αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Είναι η πιο φτωχή χώρα της Αμερικανικής Υπήρου και από τις φτωχότερες στον κόσμο, αλλά έχει υψηλό δυναμικό στο γεωργικό και τουριστικό τομέα. Το θέμα του ύδατος πρέπει να αντιμετωπιστεί Έξι χρόνια μετά το σεισμό, περίπου 80% από τα 12 εκατομμύρια, συγγνώμη, τα 12 δισεκατομμύρια που είχαμε υποσχεθεί για να ανοικοδομηθεί χώρα έχουν δαπανηθεί. Αλλά εάν κάνει κανεί μια βόλτα στη χώρα, διαπιστώνει ότι το μεγαλύτερο τμήμα αυτού του ποσού δεν έφτασε στον πληθυσμό. Αυτό αυξάνει τη δυσπιστία και έναντι των διεθνών οργανισμών, γιατί ο τρόπο παρέμβασή του έχει δημιουργήσει πολύ δυσπιστία. Δεν θα αναφέρω ονόματα. Πρέπει να του δώσουμε και πάλι ελπίδα και εμπιστοσύνη στην εκλογική διαδικασία, τα, δεσμικά όργανα, τα θεσμικά όργανα έτσι μόνο θα ξεπεράσουμε το παρόν αδιέξοδο. Τελειώνω, τελειώνω Πρόεδρε. Πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε αυτά που γίνονται στην ΑΕΤ, ιδιαίτερα μετά τι 7 Φεβρουαρίου, όταν θα πρέπει να βαρτηθεί ο κ. Μαρτέλη. Κυρία Επίτροπε, μπορείτε να βασιστείτε σε εμά. Ο διάλογο και η συνένεση είναι το καθήκον μα και θα συμβάλλουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοράο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κοιτάξτε και εγώ θα έπρεπε να έχω πάει ε, με αυτή την αποστολή που ακυρώθηκε και συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είπε ο κύριος Βαλεντσιάνο σχετικά ε, με το ότι είναι απαραίτητο να ε, λάβουν χώρα το στομό των δυνατών οι εκλογές. Τι να πει κανείς για την ΑΕΤ. Η ΑΕΤ μαστίζεται από πείνα και φτώχεια και αυτά πριν από το σεισμό και μετά το σεισμό εντάξει την πρόσεξαν τα Ηνωμένα Έθνη και Ευρώπη παρόλα αυτά εκεί υπάρχουν τα ίδια προβλήματα είναι μια ευαίσθητη δημοκρατία. Θα μπορούσαμε χωρίς ενδιασμό να πούμε ότι ο σεισμός του 2010 ήταν και εξακολουθεί να είναι ε, κάτι το οποίο εκμεταλλεύτηκαν οι πολιτικές δυνάμεις ανά, την, ε, ανά τον κόσμο γενικώ. Υπήρξε ένας νόμος για την εκμετάλλευση των πρώτων υλών από πλευράς πολυεθνικών ή αν θέλετε η αποψήλωση, οι υπερχιλήσει των ποταμών. Δυστυχώς ε, κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά τα θέματα, κανείς δεν ενδιαφέρεται να δώσει μια προοπτική βιώσιμη ανάπτυξη στη χώρα. Ε, θα ήθελα να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσον πραγματικά μπορούμε εμείς να είμαστε καθοριστικοί παράγοντες στην εξέλιξη της χώρας. Ευχαριστούμε ο κύριος Παντσέρη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας ε, στις 25 Οκτωβρίου, σήμερα στην IT βιώνουμε μια μεγάλη πολιτική αστάθεια που μπορεί να καταστρέψει αυτή την έθραυστη ε, ε, κατάσταση που υπάρχει στη χώρα. Θα πω το εξή. Η εκλογική αποστολή παρακολούθηση των εκλογών διαπίστωσε ότι υπήρχε ηρεμία κατά διάρκεια των εκλογών, καλύφθηκαν τα διεθνή στάνταρτ. Παρόλα αυτά όμως ε, εκείνοι που έχασαν ε, θέλησαν να ταράξουν τον κόσμο λέγοντας διάφορα ότι δεν ήταν σωστή η εκλογική διαδικασία. Ε, και τα μέσα ενημέρωση συνέβαλαν και αυτά στο να δημιουργήσουν εντύπωση της νοθείας των εκλογών. Εμείς όμως ήμασταν εκεί και βιώσαμε, το είδαμε μόνοι μας και με την πολύ καλή δουλειά της κυρίας Βαλεντσιάνο ότι η εκλογική διαδικασία ήταν άμεπτη. Τώρα λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα συγκεκριμένο καθήκον δηλαδή να απευθυνθεί σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, να τα καλέσει να αναλάβουν πολιτική και ηθική ευθύνη εξ του λαού για να σταματήσει ε, το ο πολιτικός αποκλεισμός και να γίνουν σεβαστά τα αποτελέσματα του Οκτωβρίου. Είναι λοιπόν απαραίτητο σύντομα να οργανωθεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα που θα βασίζεται στην επικύρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου γύρου εκλογών. Και κυρία Επίτροπε, εμείς επιθυμούμε σε αυτή τη γραμμή να παραμείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με συνέπεια και αποφασιστικότητα. Όλοι μας έχουμε το καθήκον να βοηθήσουμε την ΑΕΤ στη δημοκρατική διαδικασία που θα της εξασφαλίσει σταθερότητα και που θα της δώσει προβλήματα σε πολλά, ε, λύσεις σε πολλά προβλήματα που μαστίζουν τη χώρα, οικονομικά, κοινωνικά. Ε, πρέπει να αποκαταστήσει ζημιές που προκλήθηκαν από το σεισμό. Έχουμε ένα τεράστιο καθήκον και οφείλουμε να το ε, σεβαστούμε και να το υλοποιήσουμε μέχρι τελευταίες ρανίδος. Επόμενη μιλήτρια, κυρία Μίτσι. Ευχαριστώ. Ναι, μεν έγιναν εκλογέ στι 25 Οκτωβρίου που θεωρήθηκαν ε, σωστές εκλογές. Αλλά υπήρξαν κάποια προβλήματα και αναβλήθηκε δύο φορές ο δεύτερος γύρος. Όμως, ως παρατηρητές που ήμασταν ε, εκεί και θέλαμε να παρατηρήσουμε το δεύτερο γύρο, πρέπει να πω ότι είναι πολύ λυπηρή η κατάσταση. Λιγότερο από 48 ώρες πριν από την ε, ημερομηνία διεξαγωγής τους αναβλήθηκαν για τρίτη φορά επαόριστον ενώ υπήρχαν ε, βίες διαδηλώσεις, δολοφονίες, κτίρια και αυτοκίνητα πυρπολούντο κτλ. Η ΑΕΤ είναι από τις φτωχότερες χώρες στον κόσμο. Άρα όντως πρέπει να υπάρξει αλλαγή. Αν δεν υπάρξει αλλαγή ο κίνδυνος της αύξησης ακόμη περαιτέρω της φτώχειας είναι υπαρκτός και αυτή η φτώχεια ε, σημαίνει ότι δεν υπάρχει υγεία, δεν υπάρχει εκπαίδευση, δεν υπάρχουν υποδομές και σε όλα αυτά προσθέθηκαν βέβαια καταστροφές του καταστροφικού σεισμού του 2010. Η χώρα χρειάζεται λοιπόν απεγνωσμένα να επανακτήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών της. Η βία πρέπει να σταματήσει και οι κάτοικοι της ΑΕΤ πρέπει να έχουν τίμιε και δημοκρατικέ εκλογέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει μέσω μια ειδική αποστολή για να βοηθήσει τη διαπραγμάτευση μεταξύ των ε, πολιτικών κομμάτων για μια νέα ημερομηνία για να σταματήσει η βία και για να βοηθήσουμε για μια ταχεία επίλυση της κρίσης. Ευχαριστώ. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Κέντζε. Ενάμιση λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ την κυρία Βαλενθιάνο και όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν σε αυτή την αποστολή. Συμμετείχα στην αντιπροσωπεία της, εκλογής, της αποστολής παρατήρησης των εκλογών στις 25 Οκτωβρίου του 2015. Η Αιτή είναι μια χώρα η οποία στενάζει και προσπαθεί να ανακάμψει από τις ε, καταστροφικές, καταστροφικές συνέπειες του σεισμού που την έπληξαν ε, ε, πρόσφατα. Η χώρα ζει μέσα από μεγάλες αντιφράσεις, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά διεκδικεί το δικαίωμά τους σε ελεύθερες και δημοκρατικές εκλογές. Εμείς καταφέραμε να ε, γίνουν όντως οι εκλογές αυτές. Χάρη στην παρουσία μας στην ΑΕΤ στις 25 Οκτωβρίου έγιναν ομαλά οι εκλογές χωρίς νοθεία σε πνεύμα νομιμότητας και σεβασμό των κανόνων όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου. Ο κόσμος μας υποδέχθηκε με ενθουσιασμό και αυτό ε, κατέδειξε ότι είναι ακόμα πιο σημαντική η παρουσία μας στο νησί παρά το γεγονός ότι ήταν ισχνή η συμμετοχή στις εκλογές πρέπει να... Ε, ομολογήσω λόγω της ε, ε, μικρής εμπιστοσύνης που υπάρχει στις τοπικές, ε, ε, στις τοπικούς θεσμούς. Υπάρχουν δύο υποψήφισμοι. Θα πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν τη διαδικασία και να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας. Να διασφαλίσουμε το συντομότερο δυνατόν η ΑΕΤ να έχει δημοκρατικούς και σταθερούς θεσμούς που θα μπορέσουν να βγάλουν τη χώρα από αυτή την επισφελής θέση στην οποία βρίσκεται εδώ και πάρα πολύ καιρό πλέον. Υπενθυμίζω ότι καθήκον της αποστολής παρατήρησης των εκλογών είναι και η προαγωγή της δημοκρατίας ε, για την ειρήνη και την ασφάλεια. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε μια διαδικασία η οποία κατά την άποψή μας δεν έχει ακόμα περατωθεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα περνάμε στη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Ο κύριος Πόλτσακ καταρχάς. Ευχαριστούμε. Συμφωνούμε με αυτά τα οποία υπόθηκαν. Είναι όντως γεγονός ότι όταν προκύπτει μια θεσμική κρίση σε μια χώρα γιατί ένας υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές δεν σέβεται το αποτέλεσμα και δεν σέβεται ότι δεν αναγνωρίζει ότι οι εκλογές ήταν ε, τίμιες τότε προκύπτει πρόβλημα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να καταλήψουμε τη χώρα αυτή και τον πληθυσμό της. Θεωρώ ότι κανείς μας δεν έχει τέτοια πρόθεση φυσικά. Πρέπει να εξακολουθήσουμε, να παρακολουθούμε την κατάσταση, ίσως να στείλουμε άλλη μία αποστολή για να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές και για να υπάρξει περαιτέρω εκδημοκρατισμός. Θα ήταν λάθος πιστεύω να τα εγκαταλείψω. κύριος Μαριάς. Σαν Έλληνας Ευρωβουλευτής εκφράζω την αλληλεγγύη μου στο λαό της Αιτής τον πρώτο λαό που αναγνώρισε την ανεξαρτησία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους μετά την επανάσταση του. 1821. μετά το σεισμό του 2010 η μκο αλλά και η δύση επέβαλαν μια κυβέρνηση παρία. μάλιστα στην αϊτή συμβαίνει το παράδοξο η διεθνής κοινότητα να διαχειρίζεται εκεί δέκα φορές περισσότερα κεφάλαια από ότι ο προϋπολογισμός της αϊτής. πρόκειται για ένα φαινόμενο σύγχρονο χούλιγοντιανού δίθεν ανθρωπισμού που όμως απέτυχε πλήρως αφού εμβάθυνε την επισητιστική κρίση ξεκλήρισε τους αγρότες και απέτυχε να διοργανώσει δημοκρατικές εκλογές. γι' αυτό το λόγο έχει απέναντί του τον ίδιο τον πληθυσμό της αϊτής που έχει ξεσηκωθεί. η πορεία προς τις εκλογές χαρακτηρίστηκε από αμφισβητήσεις και βία και υπάρχει αμφισβήτηση από ό,τι ακούστηκε και για το αποτέλεσμα των εκλογών του οκτωβρίου του. 2015 ήδη υπάρχει αδιέξοδο καθώς αναβάλλονται συνεχώς ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών και το βέβαιο είναι ότι ο λαός της αιτίας θα στείλει μήνυμα με πολλούς αποδέκτες για τη δημοκρατική μετάβαση την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας και το χτύπημα της φτώχειας. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Όταν τον Ιανουάριο του 2010 η ΑΕΤ, επλήγει από αυτόν τον καταστροφικό σεισμό και είχαμε πάνω από 200.000 νεκρούς, τότε όλοι επιδείξαμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας, ξέροντας ότι ήταν από τα πιο φτωχά κράτη του κόσμου και ότι ούτως ή άλλως ακόμη και πριν το σεισμό ο πληθυσμός ζούσε σε φτώχεια, διαφθορά και αστάθεια. Ελπίζαμε όλοι ότι αυτές οι εκλογές που είχαν προβληθεί για πέρυσι και που έλαβαν χώρα με ελεύθερο και τίμιο τρόπο με βάση την αποστολή παρατηρητών συναδέλφων μας, όλοι ελπίζαμε ότι μια νέα διαδικασία σταθεροποίησης θα προέκυπτε, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη. Η Ευρώπη έχει βοηθήσει την ΑΕΤ στις πιο δύσκολες στιγμές, ήμασταν στο πλευρό τους και κατά τις τελευταίες εκλογές. Η Ευρώπη πρέπει λοιπόν να συνεχίσει την συμπαράστασή της, γιατί σίγουρα η βοήθειά μας είναι απόλυτα απαραίτητη για τον λαό. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος, λίγη διαδικασία προσέλκυσης της προσοχής του Πρόεδρου και τώρα για την ολοκλήρωση της συζήτησης έχει το λόγο η επίσημος κυρία Κρέτου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ήταν πολύ χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για τη σαφήνεια των παρεμβάσεών τους και φυσικά και για τις προσπάθειες ε, για εξέβρεση λύσης σε αυτό το αδιέξοδο το οποίο αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή στην ΑΕΤ. Βεβαίως ε, το θέμα είναι η κρίση ε, λόγω των εκλογών και είμαι βέβαιη ότι γνωρίζετε όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη στους Αιτινούς. Ε, η Αιτή είναι μία από τις ε, φτωχότερες χώρες στον κόσμο και τους παρέχει στήριξη εδώ και χρόνια τώρα. Μετά από το σεισμό του 2010, ένας στους δύο Αιτινούς έχει πληγεί από κάποια ε, ε καταστροφή και έχει λάβει βοήθεια. Ε, νομίζω όμως ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί η διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και άλλα μέσα για να υποστηρίξουμε ε, μία λύση στην Αιτή για την παρούσα κρίση που θα σέβεται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ολοκληρώσω ε, επισημένοντας για άλλη μια φορά ότι εκτιμώ το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην παρατήρηση των εκλογών και στην ε, διατήρηση αυτού του σημαντικού θέματος ε, στη διεθνή Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε.